αντιμετωπίζουμε τόσο μεγάλη ευελιξία όσο τη δική σας. Ωραία. Έληξε αυτή η συζήτηση και όπως γνωρίζετε θα ψηφίσουμε αύριο στις 11.30 την έκθεση αυτή και τις τροπολογίες της. Θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Καταρχήν να σας πω ότι λάβαμε από το Συμβούλιο δύο θέσεις για πρώτη ανάγνωση που θα πρέπει να εγκρίνουμε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής. Οι τίτλοι θα παρουσιαστούν στην ε, παρούσα Ολομέλεια, στην παρούσα Σύνοδο. Και η διαδικασία ξεκινάει από τις 26 Οκτωβρίου. Από τους πράσινους έλαβα ένα αίτημα διορισμού που ε, εντάσσεται στην παρούσα σύνοδο και εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνεται